So, liebe Kolleginnen, Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ε, αρχίσουμε. Καθίστε παρακαλώ όλοι. So, schönen guten Morgen allerseits, liebe Kolleginnen und Kollegen. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας. Ελπίζω όλοι σήμερα το πρωί και οι διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, είχατε καλές καλοκαιρινές διακοπές και ότι είσαστε πίσω με όρεξη. Κάποιοι φαντάζομαι είναι ακόμα στο δρόμο, έρχονται. Ίσως μέχρι τις 9.30 ελπίζω να είναι εδώ, γιατί τις 9.30 θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, να αρχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Να βρω κι εγώ εδώ τα χαρτιά μου. Μια στιγμή. Λοιπόν, έχουμε δύο νέους συναδέρφους που αντικαθιστούν κάποιους, τον Ζαμαρί Καβαντά και τον κύριο Πριόρης. Ελπίζω να είπα τα ονόματα λίγο πολύ καλά. Δεν τα λέω καλά. Τέλος πάντων, είναι δύσκολα τα ονόματα αυτά για μένα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε όλες τις γλώσσες σήμερα, εκτός από μαλτέζικα, κροατικά και ιρλανδικά. Έχει υπάρξει διάλογος ανάμεσα στα Ηνωμένα Έθνη και την Επιτροπή μας για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες. Ο διάλογος αυτός έλαβε χώρο 27 και 28 Αυγούστου. Ο συνάδελφός μας, ο κύριος Κόζα, συμμετείχε και εκείνο θα μας ενημερώσει, θα μας παρουσιάσει τις εξελίξεις όσον αφορά τις συζητήσεις αυτές. Παρακαλώ κύριε Κόζα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόεδρε θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα και θέλω να αρχίσω με τα γεγονότα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν υπάρχει αυτή η σύμβαση, σύμβαση για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνυπογράψει τη σύμβαση αυτή. Δεν υπογράφουμε δηλαδή αναχώρα, αλλά πρόκειται για μια ολόκληρη ομάδα χωρών, για ένα διεθνή οργανισμό. Και υπάρχει ένα σώμα το οποίο επιβλέπει πώς εφαρμόζεται η σύμβαση αυτή στην πράξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ανέλαβε αυτό το έργο. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αποφάσισαν λοιπόν να θέσουν ένα πλαίσιο για να επαληθεύσουν την ε, εφαρμογή της σύμβασης αυτής. Τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές συμμετέχουν σε αυτό το έργο. Η Επιτροπή μας έχει ηγετικό ρόλο, εγώ είμαι ο υπεύθυνο και εκτός από τη δικιά μας Επιτροπή συμμετέχει και η ΛΥΜΠΕ και η ΠΕΤΗ πολιτικών ελευθεριών και αναφορών δηλαδή. Τον Απρίλιο αρχίσαμε τις εργασίες μας και τον Απρίλιο πήγα στην Γενέβη για να συμμετάσχω εκεί σε έναν διάλογο. Εκεί εξηγήσαμε ποιο θα είναι το πλαίσιο ακριβώς και τώρα τον Αύγουστο στις 27 και 28 Αυγούστου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια παρουσίαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά έστειλε ένα ερωτηματολόγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια συγκέντρωσε τις απαντήσεις και τις πήγε στη Γενέβη. Εκεί εκπροσώπησε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση και έδωσε τις απαντήσεις μας. Η Επιτροπή Απασχόλησης θα πρέπει στο μέλλον να εργαστεί πάνω σε αυτό το θέμα. Η Επιτροπή σε θα δώσει τα συμπεράσματά της σήμερα ή αύριο και εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε. Είτε με νέες προτάσεις όσον αφορά το νομοθετικό έργο, είτε αλλιώς με άλλα έγγραφα. Τώρα, πρώτα απ' όλα, θέλω να αναφέρω τα μέτρα λιτότητας που έχουν να κάνουν βέβαια με την οικονομική κρίση στη συνέχεια στα διορθωτικά ταμεία και τη χρήση των διορθωτικών ταμείων. Ουσιαστικά πάνω σε αυτά τα θέματα πήραμε ερωτήσει. Και μετά υπήρξαν και κάποια άλλα ζητήματα, όπως το πώς η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα στηρίξει την εφαρμογή της προσβασιμότητας των ατόμων αυτών στην εργασία. Όπως γνωρίζουν και οι συναδελφοί, πριν από τέσσερα χρόνια η Επιτροπή μας υποσχέθηκε ότι θα επιμείνει για νέες προτάσεις όσον αφορά την ε, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες. Εκπροσωπούμε λοιπόν τους ανθρώπους που ζουν με αναπηρίες για να δούμε κατά πόσο υπάρχει περιορισμό στα δικαιώματά τους, είτε πρόκειται τα δικαιώματά τους στο εκλέγει και εκλέγεστε, είτε σε άλλα πράγματα. Αναφέρθηκε ας πούμε η άδεια μητρότητας ή άλλα ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ρωτήθηκε για πάρα πολλά από αυτά τα ζητήματα. Και το τελευταίο στο οποίο θα αναφερθώ είναι το πλαίσιό μας. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο δουλεύουμε είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως συμμετέχει σε αυτό το πλαίσιο. Θα έλεγα ότι η Επιτροπή της Γενέβης θα μας επικρίνει εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Τώρα, εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς ε, μιλήσαμε για το ψήφισμα που εγκρίναμε τον Μάιο στην Ολομέλειά μας. Ήταν κάτι πολύ θετικό, ένα πολύ θετικό βήμα. Οι συνάδελφοι ήδη γνωρίζουν ότι το φθινόπωρο θα υπάρξει μια νέα έκθεση που συντάσσεται για την εφαρμογή της σύμβασης αυτής των Ηνωμένων Εθνών. Και όλα αυτά δείχνουν ότι η Επιτροπή Απασχόλησης πραγματικά έχει αναλάβει τη δέσμευση, την υποχρέωση να δουλέψει πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και θέλω να σας υπενθυμίσω και κάτι. Το Σεπτέμβριο δημιουργήθηκε ένα δίκτυο στο Κοινοβούλιο με νέα κοινοβουλευτικέ επιτροπές που έστειλαν μέλη στο δίκτυο αυτό, σε αυτή την ομάδα και νομίζω ότι η δουλειά μας είναι πραγματικά δουλειά ποιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο για να σας ενημερώσω για όλα αυτά. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κύριε Κώσα. Σύντομη αλλά περιεκτική η ανάπτυξη του θέματος από σας. Τρίτο θέμα τώρα, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης, πρόσβαση εργαζόμενων σε υπηρεσίες κινητικότητας και ενοποίηση αγορών εργασίας. Στις 23 Έκτου είχαμε ψηφίσει την έκθεση του κ. Μπέκερ. Στο μεταξύ έχουν διεξαχθεί, γιατί είχαμε δώσει τότε και τη διαπραγματευτική εντολή βέβαια, έχουν διεξαχθεί συνομιλίες με το Συμβούλιο πρώτη συνάντηση έγινε στις 15 ε, Εβδόμου, διεξήχθη με επιτυχία, έχουν γίνει διαπραγματεύσεις για τις πρώτες παραγράφους του κειμένου, επιτεύθηκαν πρόοδοι, εδώ αυτό μου έχουν σημειώσει, δεν θέλω όμως να προκαταλάβω τα όσα θα πει ο ίδιος ο κύριος Μπέκερ. Περιοριστείτε σε 10 λεπτά για να προλάβουμε να ψηφίσουμε. Κύριε Μπέκερ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που σας βλέπω στην Προεδρία και εκφράζω προσωπικά δηλαδή την ικανοποίησή μου που είστε ξανά στον θόκο του Προέδρου. Χθες έγινε ο δεύτερος τριμερής διάλογος. Έχουμε συμφωνήσει επί της διαδικασίας με την έννοια ότι θα συζητήσουμε πρώτα τα άρθρα και κατόπιν τα εκτιμώντας. Στα άρθρα έχουμε προχωρήσει αρκετά αφενός για το πώς θα δημιουργηθεί το δίκτυο ΕΟΡΕΣ, γιατί υπάρχουν διαφορετικά, διαφορετικές δομές. Υπάρχει Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού, Εθνικά Γραφεία Συντονισμού, υπάρχει το ερώτημα του προτιμησιακού ρόλου των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, τίθεται ξανά και ξανά το θέμα των ιδιωτικών παρόχων, των διαφόρων μη κρατικών οργανώσεων. Όλα αυτά είναι αρκετά περίπλοκα. Πάντως έχουμε προχωρήσει στο βαθμό που να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε συμφωνήσει επί κάποιων αρχών, θα συζητηθούν ακόμη κάποιες διατυπώσεις. Υπάρχει μια πτυχή που έχει σημασία για μας, να καθοριστεί δηλαδή ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Δεν πρόκειται για αντίφαση, πρόκειται για τεχνικά θέματα περισσότερο. Νομίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε βήμα-βήμα όπως έχουμε ήδη καθορίσει εδώ στην Επιτροπή Απασχολήσεως. Γεγονός είναι και είναι ικανοποιητικό ότι είναι θετική, επικοδομητική ατμόσφαιρα και από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς συναισθηματικούς φραγμούς. Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως και την πρόεδρό μας και βεβαίως τα πρόσωπα της γραμματείας. Μπάρμπαρα και άλλοι που η βοήθειά τους είναι ανεκτήμητη. Το ίδιο ο νομικός μας σύμβουλος Μάριο, ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Ιδιαίτερα όμως τονίζω την συνεργασία με τους σκιώδεις συγητές και τους συνεργάτες του. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ. Ο Χέντελ. Καλά μου φαίνονται όλα αυτά και εύχομαι καλή επιτυχία στις περαιτέρω συζητήσεις σας. Μάλλον μου φαίνεται ότι τώρα βιαστήκαμε κάπως γιατί η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 9 και 30. Ε, νομίζω ότι παραπάτησα τον γκάζι, άρα θα χρειαστεί να κάνω μια, ένα μικρό διάλειμμα. Είμαι βέβαιος ότι θα θέλετε όλοι να πείτε τι κάνατε στις διακοπές στους διπλανούς σας, οπότε ε, λίγο διάλειμμα δεν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 Κυρίες και κύριοι, ας προχωρήσουμε τότε στην ημερήσια διάταξη, ε, στην ψηφοφορία δηλαδή για τον προϋπολογισμό, τουλάχιστον το τμήμα εκείνο το οποίο μας πέφτει ως ε, Επιτροπή Απασχολήσεως. Έχουμε συνολικά 94 τροπολογίες Και αρχίζουμε αμέσως την ψυχοφορία Και πρώτη... Πρώτη 62-38. Παρακαλώ ψήφι υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 62-32. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62-39 υπέρ κατά απορρίπτεται 62-45 κατά εγκρίνεται 62-00 υπέρ κατά Το πρώτο κερδίζει. Ευχαριστώ. Αν θέλετε επαλήθευση. Καλά λοιπόν. 62-0-0. Ψηφίσατε. Τέλος. 22 υπέρ 17 κατά. Η επόμενη εκπίπτει. 62-46 λέει ο πρόεδρος τώρα. ψηφιπέρ Κατά. False, false λένε οι διάφοροι. Εκπίπτει λοιπόν. λοιπόν. 46 εγώ εξεφώνησα λέω. Ξαναλέω λοιπόν 62-46 υπέρ κατά απορρίπτεται 62-40 υπέρ κατά εγκρίνεται 62-01 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. 62-02 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62-33 υπέρ. Κατά. Το πρώτο κερδίζει, εγκρίνεται. 62-42 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 62-43 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση παρακαλώ. 62-43. Ψηφίσατε. Εγκρίνεται. 62-48 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 62-49 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 62-34 υπέρ κατά εγκρίνεται αυτή 62-50 υπέρ κατά απορρίπτεται σαφώς 62-03 υπέρ κατά εγκρίνεται και άρα εκπίπτει 6251 και 6252. Άρα 6235 τώρα υπέρ κατά εγκρίνεται 6253 και 54 είναι ταυτόσιμες άρα μαζί υπέρ κατά απορρίπτονται. Α, θέλετε τσεκ. Καλά λοιπόν. 62, 53 και 54. Εσείς είναι σούπερ. Έχουμε εδώ δίπλα μας ένα μέλος, έχω μάλλον δίπλα με το ένα μέλος, που δεν έχει την κάρτα της. Να σημειώνετε την ψήφο. Ναι, ναι, θα ε, κάνουμε τότε με το χέρι. Παρακαλούμε τότε να δείχνετε καθαρά με το χέρι, ναι, όχι κλπ. Μόλις βλέπω ότι οι σοσιαλδημοκράτες έχουν μια ψήφο παραπάνω, ποιος θα αποχωρήσει και ο θελός, ή θα αποφασίσει η Σιγιούτα. Γιούτα παίζεις με ένα παίχτη παραπάνω. Ωραία, εντάξει, τώρα είμαστε εντάξει. Άλλο τίποτε υπάρχει. Όχι, εντάξει. Ωραία, τώρα είμαστε σωστά στα νούμερα και το αποτέλεσμα ...62, 53 και 54 εγκρίνονται λοιπόν με μία ψήφο διαφορά. 62-55 υπέρ κατά Α, με συγχωρείτε λέει. Είμαστε τώρα στην 62-56. Μόνο στα σχόλια, Ρημάξε Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 62.05 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 62.57 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 62.58 υπέρ, κατά. Εδώ χρειάζεται επαλήθευση 6258. Πάλι μια παραπάνω ψήφος στους σοσιαλδημοκράτες. Τώρα είναι εντάξει. 62-58 έχει στο μεταξύ εγκριθεί. 62-60 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 62-60 τα σχόλια τώρα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 62-62 υπέρ. Κατά. Κάπως ασαφές το αποτέλεσμα. Ας το ξαναδούμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Εγκρίνεται. Σαφέστατο βέβαια. 62-07 υπέρ. Κατά. Δύσκολο να πει κανείς, σας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση πάλι. Ψηφίσατε. Απερίφθη. 62-63 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται σαφώς. 62-64 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται και αυτή. Τώρα 62-64 remarks. Σχόλια. Υπέρ. Εγκρίνεται.

Απορρίπτεται αυτή. 62-67 υπέρ. Κατά. Και αυτή απορρίπτεται. 62-67 τα σχόλια υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 62-68 υπέρ κατά εγκρίνεται 62-69 υπέρ κατά εγκρίνεται 62-70 είναι ταυτόσιμη. χρειάζεται να ψηφιστεί ξεχωριστά δεν χρειάζεται όχι 62-71 υπέρ 62-72 υπέρ κατά στην λίστα της ψηφοφορίας υπάρχει ένα λάθος. Κατά τα όσα μου λένε το 6271 θα έπρεπε να εκπίπτει εφόσον εγκριθούν τα προηγούμενα 6269 και 70. Σωστά το είπα. Ωραία. Ωραία λοιπόν τώρα. Ξεκαθαρίστηκε. Τώρα όμως 6272. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Σαράντα υπέρ εννέα κατά. Μου φαίνεται ότι δεν βλέπω καλά σήμερα. Τώρα είμαστε στην 62.08 υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση? Όχι. Όχι, εντάξει. Εξήντα δύο υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Εξήντα δύο κατά εγκρίνεται και αυτή 6279 υπέρ κατά νομίζω ότι υπερτερούν τα υπέρ 6210 υπέρ κατά απορρίπτεται αυτή 6280 υπέρ κατά απορρίπτεται τσεκ οκ 62-80 επαλήθευση ψηφίσατε απορρίπτεται όπως δείχνει το αποτέλεσμα 62-11 υπέρ κατά εποχης απορριπτεται απορρίπτεται 62-81 υπέρ κατά απορρίπτεται 62-12 υπέρ κατά απορρίπτεται 62-82 υπέρ κατά επαλήθευση Ψηφίσατε. Απερίφθη. 62-13 υπέρ. Κατά. Υπερτερούν τα όχι, αλλά απορρίπτεται. 62-83 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. ...62-84... ...πρώτα οι αριθμοί... ...υπέρ... ...κατά... ...απορρίπτονται... ...62-84... ...τα σχόλια... ...υπέρ... ...κατά... ...απορρίπτεται... Οκ, okay, επαλήθευση 6284 remarks. Ψηφίσατε. Το αποτέλεσμα. Απερίφθη. 62-85 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 62-15 υπέρ κατά απορρίπτεται 62-16 υπέρ κατά εγκρίνεται 62-17 υπέρ κατά Ας κάνουμε μια παρήθευση 62-17 σαφές το αποτέλεσμα. Το λέω χωρίς απολύτως καμιά πολιτική αξιολόγηση. Σας παρακαλώ σηκώνετε ψηλά τα χέρια για να σας βλέπω και αυτό το λέω για τους συντηρητικούς τώρα. 6286 υπέρ. Κατά. νομίζω ότι υπερτερεί το δεύτερο, άρα απορρίπτεται. 62-18 υπέρ κατά. Εξήντα δύο Σαφώς απορρίπτεται. Μήπως σας φαίνομαι ότι πάω πολύ γρήγορα και γι' αυτό μπερδεύεστε με τα χέρια πάνω κάτω. Δεν καταλαβαίνω τελικά πώς είναι υπέρ και πώς κατά. Έτσι όπως γίνεται. Σας παρακαλώ να μην διαμαρτύρεστε. Νομίζω ότι τα πάτε θαυμάσια αλλά όταν οι δυο συντονιστές μας που κάθονται εκεί μπροστά των δύο μεγάλων κομμάτων ψηφίζουν με τον ίδιο τρόπο, εγώ νομίζω ότι τα πάτε πολύ καλά. Σκέπτομαι μόνο ότι ίσως θα μπορούσατε να επιταχύνετε γιατί αν έχουμε πολύ περισσότερες τροπολογίες κάποια στιγμή θα χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο. Σημειώνω πολύ προσεκτικά αυτό που είπατε και σας βεβαιώνω ότι μπορώ και πολύ πιο γρήγορα. 62-87 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 62-19 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 62-20 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 62-21 υπέρ. Κατά. λίγο δύσκολο. Επαλήθευση. 62-21 επαλήθευση. Ψηφίσατε. Αποτέλεσμα. Μάλιστα. Μικρή, πολύ μικρή διαφορά. Ακόμα και αν προσθέσουμε την ψήφο σας ε, είναι ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. 62-22 υπέρ, κατά, Η κατάσταση διαμορφώνεται με παρόμοιο τρόπο. 62, 22 ηλεκτρονικά. Τέλος, ισοψηφία. Απορρίπτεται. Α, να συνυπολογίσουμε και την ψήφο σας, άρα τότε το αποτέλεσμα είναι 25-24, άρα υπερψηφίζεται, εγκρίνεται. Διακόπτει ο πρόεδρος. Ορίστε. Ναι. Οκ, συμβαστικη 62.95. Υπέρ, κατά. εγκρινεται 62.24. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 62-25 υπέρ, κατά, Νομίζω ότι εγκρίνεται. Θέλετε παρήθευση οπωσδήποτε. Καλά λοιπόν. 62-25. Check. Ψηφίσατε. Απερίφθη. 62-26 υπέρ κατά απορρίπτεται 62-27 υπέρ κατά απορρίπτεται 62-89 υπέρ κατά εγκρίνεται 62-28 υπέρ Α, εκπίπτει τούτη εδώ. Άρα, συμβαστική 62-94. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 62-91 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 62-30 υπέρ. Κατά. και αυτή. 62-92. Δηλαδή οι του αριθμού υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 62-92 τα σχόλια υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 62-31 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 62 93 υπέρ κατά εγκρίνεται τελική ψηφοφορία δεν γίνεται τα διαβιβάζουμε τα αποτελέσματα αυτά στην αρμόδια επί επιτροπή όπως άλλωστε εγκρίναμε σήμερα Λίγη σήμερα η ημερήσια διάταξη της ε, Επιτροπής Απασχολήσεως. Σας ευχαριστώ όλους και όλους και θα τα ξαναπούμε στις 15 Ενάτου. Από τις 9.30 και 30 έως τις 12 και 30 και επίσης το απόγευμα στα γνωστά ωράρια.